Η συμφωνία Μερκοσούρ εμπεριέχει στεναρά κεφάλαια περί αναπτύξης και εμπορίου. Ε, συμμορφώνεται αυτό το τμήμα με ύψιστε προδιαγραφέ όπω άλλε συμφωνίε, όπω η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ιαπωνία ή το εμπορικό τμήμα τη Γενική Συμφωνία με το Μεξικό. Η συμφωνία του Μερκοσούρ περιέχει συγκεκριμένο άρθρο περί αλλαγής κλίματος και δεσμεύει τα συμβαλόμενα μέρη ενεργά να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης υπήρχαν δεσμεύσει για την καταπολέμηση της αποδάσωσης, πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα ενισχύουν αυτές οι υποχρεώσεις. Παραδείγματο χάρη να μην ε, πωλείτε, να μην αγοράσετε κρέα από κτηνοτροφικέ μονάδε που ε, δημιουργούνται σε περιοχέ αποδασωμένε πρόσφατα. Εμπεριέχονται άλλε υποχρεώσει όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Διαφυλάσσει σχετικέ πρωτοβουλίε για βιώσιμη γεωργία. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η δράση ιδιωτικού τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μηδενική αποδάσωση όσον αφορά τον τομέα αυτό και πρωτοβουλίε για το πάγωμα ε, παραγωγή σόγιας στην Βραζιλία, ούτω ώστε να μην γίνεται η επέκταση των ε, σοδιών αυτών ει βάρο των δάσων. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουμε θεματικά θέματα για πτυχέ εμπορικής φύσεω για φυσικούς πόρους, όπως είναι η βιοπικιλότητα, τα δάση, η αλληλεία, και η καταπολέμηση τη παράνομη υλοτομία. Αυτή η συμφωνία προβλέπει μια πλατφόρμα τόσο σε ενεργά να συνομιλήσουμε τι χώρε Μερκοσούρ για θέματα βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμφωνία περιγράφει διάφορους τομεί ενδεχόμενη συνεργασία, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται ότι το εμπόριο θα στηρίζει το θεματολόγιο τη βιωσιμότητας. Προσφέρει και στην κοινωνία των πολιτών και σχετικέ οργανώσει ενεργό ρόλο, ούτω ώστε να ελέγχουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων ή ονδήποτε ανησυχιών για το περιβάλλον. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, τα κεφάλαια περιμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης είναι νομικώς δεσμευτικά και εφαρμοστέα. Υπόκεινται σε συγκεκριμένου μηχανισμούς διευθετής των διαφορών και δυνατότητα καταγγελίας για μη συμμόρφωση καλύπτεται από συζητήσει μεταξύ κυβερνήσεων. Αν δεν επιληφθεί το πρόβλημα, τότε ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων μπορεί να επιληφθεί για να εξετάσει το θέμα και να προτείνει συστάσει. Η έκθεση και οι συστάσει θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται από εμπλεκόμενου φορεί καθώ και από σχετικού θεσμού των συμβαλωμένων μερών. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά θα θέλατε ισχυρότερο μηχανισμό επιβολής των μέτρων, ακόμα και με επιβολή κυρώσεων. Αυτό το θέμα συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο καθώς και στο Συμβούλιο. Επ' αυτής της βάσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε ένα σχέδιο με 15 σημεία ώστε τα κεφάλαια για αύξηση ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενώσης να είναι πιο στεναρά και πιο αποτελεσματικά και στην περίπτωση Όπω και στην περίπτωση επίλυση διμερού διαφωνία με την Κορέα, βλέπουμε ότι αυτά δεν είναι κενά λόγια. Τι πετύχαμε από το Μέρκοσουρ όσον αφορά περιβαλλοντικέ πτυχέ και πτυχέ βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά που πετύχαμε είναι αποτέλεσμα σκληρών και μακροχρονίων διαπραγματεύσεων. Αυτέ οι υποχρεώσει αποτελούν πρόκληση για τι χώρε Μέρκοσουρ, αλλά είναι έτοιμε να επομιστούν τι ευθύνε του. Μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία με το Mercosur που συμβάλλει στο βιώσιμο εμπόριο με την περιοχή συμπεριλαμβανομένων και δεσμεύσεων από τι χώρε Μερκοσούρ να εφαρμόσουν τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, θα παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον κατάλληλο μοχλό για να επιδιώξουμε του φιλόδοξου στόχου μα για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρόσφατε δασικέ πυρκαγιέ στην περιοχή του Αμαζονίου δείχνουν τα προβλήματα όσον αφορά τη βιωσιμότητα που αντιμετωπίζει το Μερκοσούρ. Αλλά, κυρία Πρόεδρε, είμαι πεπισμένη ότι αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο συνεργασία με το Μερκοσούρ. Μπορούμε να πετύχουμε την παγκόσμια μεταμόρφωση που τόσο πολύ επιθυμούμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον Επίτροπε κύριε Χόγκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να ε, εισφέρω σε αυτή τη συζήτηση και χαιρετίζω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια συζήτηση η οποία παρουσιάζει το σχέδιο του Green Deal της Επιτροπής της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Το Ευρωπαϊκό Green Deal παρουσιάστηκε εδώ την περασμένη εβδομάδα και είναι μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προαχθεί η ευημερία των πολιτών και του πλανήτη μετασχηματίζοντας το οικονομικό μας μοντέλο. Ε, είναι φιλόδοξος ο, ρόλος της, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050 ε, προστατεύοντας το κλίμα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και των πολιτών. Ε, το ενεργειακό μείγμα, οι βιομηχανικές διαδικασίες, ε, το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ενέχονται σε αυτή την αλλαγή και θα πρέπει η πολιτική να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Ε, ε, πρόκειται αυτό να συμβεί σε μονομερές και πολυμερές επίπεδο. Οι φυστάμενες συμφωνίες στο, ε, στον ΠΟΕ καθώς και οι διμερείς συμφωνίες θα παίξουν εδώ καθοριστικό ρόλο. Πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να εισβάλλει στην εφαρμογή του Green Deal. Ε, σαν κάποιο ο οποίο συμμετείχε στην διαπραγματεύσει, μπορώ να πω ότι αυτό είναι εφικτό. Οι συμφωνίε της Ευρωπαϊκή Ένωση και Μπορείου θα περιλαμβάνουν κεφάλαια βιώσιμου και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να ε, συμβάλλουμε στη σύσχεση των σχέσεων με τις χώρες των ε, Μερκοσουρ, ε, σύμφωνα με τους στόχους των Παρισίων. Και έτσι καλύπτονται, και αυτό αφορά και τις υποσχέσεις της Βραζιλίας, να αποκαταστήσει και να αναδασώσει χιλιάδες εκτάρια ε, και να θέσει ένα τέρμα σε παράνομες ε, πρακτικές αναδάσεις. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Ε, επίσης, θέματα όπως η βιοπικιλότητα συμπεριλαμβάνονται, η διαχείριση των αποβλήτων και η αλυσίδα διάθεση των προϊόντων. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των δύο πλευρών να λάβουν μέτρα και να βασίσουν την νομοθεσία στην αρχή της πρόληψης. Ε, είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά σε μια συμφωνία με ένα μείζον εξαγωγικό μπλοκ. Η συμφωνία γι' αυτό θα βοηθήσει τους ε, καταναλωτές και θα παράσχει ε, δικλείδες ασφαλείας και δικλείδες υψηλών προδιαγραφών για το περιβάλλον βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και την Συμφωνία των Παρισίων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων και προκειμένου να υπάρξουν διατάξεις για το διάλογο και θέματα συνεργασίας στους ωκεανούς, στις θάλασσες και στο θέμα της ενέργειας. Και με τον τρόπο αυτό ε, δίδονται, παρέχονται εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σήμερα δεν διαθέτει στη σχέση με τις χώρες του Μερκοσούρ. Η συμφωνία με τη Μερκοσούρ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ε, του Green Deal με άλλο τρόπο. Ε, πολλά η συμφωνία θα βοηθήσει να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα, να υπάρχουν βιώσιμες ε, πρακτικές ε, ε, προμήθειας των προϊόντων σύμφωνα με την πράσινη τεχνολογία. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ε, και αυτό θα επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών και στι τρίτε χώρε να καθαστήσουν τι κυβερνήσει του υπεόλογε εκπρόσωπου εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η εφαρμογή βεβαίω παίζει ρόλο κλειδί και θα πρέπει να έχουμε μια να ευθυγραμμιστούμε με το σχέδιο δράσης το οποίο συμφωνήθηκε τον ε, Φεβρουάριο. Η Κομισιόν θα παραμείνει γρηγόρη όσον αφορά την εφαρμογή ε, της συμφωνίας ε, και γιατί αυτό ε, ε, παίζει όλο όσο ε, αφορά τα θέματα της βιωσιμότητας του εμπορίου. Το συμπέρασμά μου είναι ξεκάθαρο, κυρία Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ όχι μόνο μπορεί να εισφέρει, αλλά είναι ουσιαστικό στοιχείο κάθε διεθνούς συμφωνίας προκειμένου να υποστηριχθεί το Green Deal. Ευχαριστώ οι πολιτικές ομάδες. Τώρα, καταρχήν, Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα, ο κύριος Σίμων. Δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ε, τα πράσινα θέματα, κατά πόσο πρόκειται για τη συμφωνία της Μερκοσούρ και κατά πόσο είναι συμβατή με το Green Deal, ε, η απάντηση είναι ναι. Μάλιστα η συμφωνία είναι μια αναγκαία συνεισφορά στον Green Deal, ακριβώ όπω το διατυπώσε και η Επίτροπο. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην ιστορία του δικαίου, γιατί και αυτό το είπε ο Επίτροπο κ. Χόγκαν, για πρώτη φορά έχουμε ένα μηχανισμό εφαρμογή σε μια πολυμερή συμφωνία υπέρ του περιβάλλοντο και των κοινωνικών προδιαγραφών. Θα διατυπωθούν κάποιε προδιαγραφέ, οι οποίε δεν θα ήταν υπαρκτέ χωρί τη συμφωνία αυτή. Γι' αυτό το ερώτημα του τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε υπερψηφίσει τη συμφωνία. Βεβαίω θα υπήρχε και τότε εμπόριο μόνο χωρί προδιαγραφέ, χωρί κανόνε. Με τη συμφωνία αυτά, αυτή πάμε, α, κάνουμε το βήμα από το μη ρυθμισμένο εμπόριο προς ένα θεμητό εμπόριο βάσει κανόνων. Κυρίες και κύριοι, ε, θα ασκήσουμε επιρροή στον κόσμο μόνο εφόσον μπορούμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία. Το είδαμε το καλοκαίρι. Ήδη πριν από θέση ισχύ η συμφωνία άσκησε πολιτική πίεση στις ε, πυρκαγιές ε, στα δάση των Αμαζονίων και με τον τρόπο αυτό προστατεύθηκαν κάποιες, φυσικές, κάποιες περιοχές. και στο παρελθόν δόθηκαν υποσχέσεις αλλά τίποτα δεν εφαρμόστηκε και έχει έρθει το... η κατάλληλη στιγμή να μην ε, λέγονται μισές ε, αλήθειες στους πολίτες. Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος πέρα από τα όρια μιας ε, απλά συμβολικής εξαγγελίας δεν θα πρέπει εμείς Ευρωπαίοι μόνο να πάμε μπροστά αλλά να φροντίσουμε τους ώστε ο υπόλοιπο κόσμος να εφαρμόσει τις δικές μας προδιαγραφές και αυτή η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα, ε, σημαντικό κομμάτι. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών τώρα για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Φαν Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ακούσαμε ήδη, η Ευρώπη βρίσκεται στην αρχή μιας νέας εποχής και με την Πράσινη Συμφωνία θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα μέλλον περισσότερο δίκαιο, περισσότερο βιώσιμο που να μην καταστρέφει το κλίμα. Ε, Συγχρόνω, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε αντιμέτωποι με μία κόπ στη Μαδρίτη που δεν ήταν επιτυχής. Ας λέμε την αλήθεια. Και ναι, μεν ήμασταν υπεύθυνοι κυρίως, ήταν η Βραζιλία για αυτήν την ας πούμε αποτυχία ή τέλος πάντων την έλλειψη επιτυχίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Να είμαστε ειλικρινεί από την αρχή. Είναι αδιανόητο οι αγρότες μας, οι μεταπιτές μας να πρέπει να κάνουν τεράστιες συμφωνίες για αυτή τη νέα πράσινη συμφωνία και από την άλλη μεριά οι εμπορικές συμφωνίες να παραμένουν ίδιες. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις αγορές μας σε αυτές τις χώρες οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν από τον κοινωνικό ανταγωνισμό προς τα κάτω, με προδιαγραφές προς τα κάτω. Και θέλω να το πω και άτυπα αλλά και επίσημα. Σήμερα δεν πιστεύω ότι υπάρχει ε, πλειοψηφία ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περάσει συμφωνία Μερκοσούρ ως έχει. Και εντάξει, μπορεί να μην έχω την απόδειξη, αλλά έχω κάποια εμπειρία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σα υπογραμμίσω λοιπόν και θα σα πω ότι είναι σημαντικό για του σοσιαλδημοκράτε να γίνεται επόμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε και ισχύει για άλλε χώρε, αλλά η Βραζιλία κυρίω, να ακολουθήσει μία στάση στι διεθνεί προδιαγραφέ. Αν θέλουν να είναι εταίροι μα, πρέπει να είναι εταίροι μα και στα μέτρα αυτά που παίρνουμε για το κλίμα. Δεύτερον, θέλουμε ε, κοινοποίηση εκ των προτέρων. Θέλουμε να αλλάξουν οι πολιτικές ε, στην Βραζιλία όσον αφορά ε, τον Αμαζόνιο. Και τώρα θέλω, και εδώ στρέφομαι στο Συμβούλιο, αλλά βέβαια και στην Επιτροπή, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και καιρό ζητάμε τα κεφάλαια για τις κοινωνικές προδιαγραφές αντιντάμπινγκ και τα λοιπά να γίνουν πιο δεσμευτικά και να προβλέπουν και κυρώσεις. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να έχουμε τέτοιες ρυθμίσεις. Το χαρτί πάει χαμένο. Λιγότερα γραπτά και περισσότερη δράση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρου της Ρινιού το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Κάνιας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ και συζητάμε για τη συμβατότητα της συμφωνίας μερκοσούρ με την Πράσινη Συμφωνία και δεν συζητάμε για την ίδια συμβατότητα που αφορά και άλλες εμπορικές συμφωνίες. Γιατί. Γιατί Κάποιοι έχουν ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση προσπαθώντα να βρούνε κάποιο εχθρόν, προσπαθώντα ε, να βρούνε μια νέα σέτα και τη βρήκανε τώρα ε, στο πρόσωπο τη Μερκοσούρ. Να είμαστε ξεκάθαροι. Η πρόεδρο Φοντερ Λέιεν, όταν μα παρουσίασε την ε, Πράσινη Συμφωνία, είπε ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να χρησιμεύσει για συνεργασία μα με του εταίρου μα για δράση υπέρ του κλίματο και του περιβάλλοντο έτσι όπως προβλέπονται από τη Συμφωνία των Παρισίων που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο κάθε διεθνούς συμφωνίας. Οπότε υπάρχει τέτοιο στόχο σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Ε, συνάδει με τη συμφωνία του Παρισιού. Ναι. Έχουν επικυρώσει χώρε Μερκοσούρ τη συμφωνία του Παρισιού και έχουν δεσμευτεί να την εφαρμόσουν. Ναι. Λοιπόν, με όλα αυτά τα ναι, τότε γιατί υπάρχει τέτοια ζήλια, επικρίσεις ε, και τόσα φοβερά πράγματα που θυμίζουν αποκάλυψη που λένε οι συνάδελφοι. Αν θέλουμε ο αγώνα μα για το κλίμα να έχει κάποιε επιπτώσει θετικέ, πρέπει να έχουμε συμμάχου. Και αυτό θα γίνει βάσει συμφωνιών. Και αυτή η συμφωνία είναι η πιο σύγχρονη από όσε έχουμε εκπονήσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως οι διάφοροι ε, λαϊκιστές βέβαια που μιλάνε κατά, αλλά εμείς χρειαζόμαστε εδώ πέρα συμφωνίες και δεσμεύσεις. Αυτή η συμφωνία πηγαίνει πιο μακριά από τα εμπορικά. Πρόκειται για μια συμφωνία που έχουν υπογράψει σύμμαχοι και τέρι, οι οποίοι πιστεύουν στην ίδια δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και πιστεύουν σε ένα πολυμερές ε, σύστημα με ε, ρυθμίσεις. Οπότε θα, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να ζούσουν όπως εμείς και μαζί μας. Οπότε η συμφωνία αυτή με την Μερκασόρ διασφαλίζει κάποιε εμπορικέ σχέσει που ήδη υπάρχουν, αλλά με κάποιε δεσμεύσει αδιαφυσβήστητε και με υποχρεώσει πολύ συγκεκριμένε. Και για όλα αυτά, και παρότι ότι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση από αυτού που πάντα είναι κατά οποιασδήποτε συμφωνία με την στήριξη άλλων οι οποίοι θέλουν να κουκλώσουν δικά του εθνικά προβλήματα και κάνουν ότι τα ξέρουν όλα εγώ σας λέω ότι βασίζονται σε παραπληροφόρηση, σε προκαταλήψει, σε ψέματα και σε όλα αυτά μαζί. Αλλά το κατά πόσο είναι συμβατή με την Πράσινη Συμφωνία, Συμφωνία Μερκοσούρη ή όχι, εγώ λέω και βροντοφωνάζω πως ναι. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων για τρία λεπτά. Η κυρία Καβατσίνη έχει το λόγο. Η Κομισιόν ε, είπε ότι το Green Deal είναι το κεντρικό της πρόγραμμα τα προσεχή έτη. Ε, και χαιρετίζω αυτή την εξεγγελία. Και με αυτό η Κομισιόν δεν απευθύνεται μόνο στην κλιματική κρίση, αλλά θέλει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα των δεκάδων χιλιάδων νέων που έχουν κατέβει στην Ευρώπη στους δρόμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι το 2050 ε, κλιματικά ουδέτερη, μας είπε η κυρία Φόντερ Λάιν. Αλλά θα ήθελα άμεσα να σας ρωτήσω το εξή κύριε Χόγκαν. Πώς συμβιβάζεται η δήλωση αυτή με την ε, παρούσα πολιτική εμπορία γιατί αν δούμε το, τη συμφωνία Μερκοσούρ, υπονομεύει όλες μας τις κλιματικές προσπάθειες. Αφορά ε, τα προϊόντα κρέατος ε, και γάλακτος. Θα γίνει η εισαγωγή της σόγια ακόμα φθηνότερη και πρόκειται προϊόντα τα οποία κάπου ε, θα πρέπει να καλλιεργηθούν. 20% της περιοχής του Αμαζονίου έχουν καεί. Το ποσοστό αναδάσωσης στη Βραζιλία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και στις περιοχές αυτές, και αυτό έγινε μόνο και μόνο για να καλλιεργηθούν ε, στα χωράφια αυτά, στις περιοχές αυτές ε, σόγια, κρέας κλπ. Ε, με τον τρόπο αυτό απειλείται από κατάρρευση ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση το προωθεί αυτό με την πολιτική εμπορίου και ε, κάνει συμφωνίες με τον Πολσονάρο ο οποίος ε, υπονομεύει, σαμποτάρει όλες τις ε, κλιματικές συμφωνίες για παράδειγμα αυτή της Μαδρίτης προκειμένου να περιοριστεί η χρήση φυτοφαρμάκων και προκειμένου να προστατευτούν τα δάση ε, θα έπρεπε να γίνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο επιτυχάνεται με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Ε, θα πρέπει να ανασταθεί εντελώ η πολιτική εμπορίου. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή ε, θα πρέπει να παλέψουμε μια διαφορετική συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ. Ε, χρειαζόμαστε βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Και εδώ θα πρέπει η Κομισιόν να μας δώσει ένα σχετικό νομοσχέδιο. Οι, Ευρω... Ε, οι χώρες μέλη θα πρέπει να μπορούν να προσαχθούν στη δικαιοσύνη λόγω εφόσον δεν ακολουθούν αυτή την πολιτική. Χρειαζόμαστε να κατοχυρηθεί η κλιματική πολιτική σε όλα τα κεφάλαια της Συμφωνίας Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη ομάδα Δαυτότητα και Δημοκρατία για δύο λεπτά, ο κ. Μπουκχάιτ έχει το λόγο στο ID. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η Συμφωνία Μερκοσούρ θα μπορούσε να είναι μια πετυχημένη ιστορία. 35 ε, τελωνικών δασμών για προϊόντα της ε, Βραζιλίας ήταν τεράστιο εμπόδιο στο εμπόριο. Ε, στη συνέχεια δεν είχαμε μόνο μία νέα υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, αλλά μία και φτιάχτηκε μία εντελώς καινούρια συμφωνία Mercosur. Ε, τι θέλουμε να εξάγουμε. Κανείς δεν... Οι χώρες της Μερκοσούρ, όσον αφορά τη αγοραστική τους δύναμη, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικά ε, αυτοκίνητα σαν αυτά που ετοιμάζονται να ξεχυθούν στους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης. Ε, τι γίνεται με το Green Deal οι επιχειρηματίε μας με τις έδρες παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι απολύτως ε, εκτεθειμένες. Οι εμπορικοί μας εταίροι όμως μπορούν να αναζητήσουν καινούριου εταίρους και στη χειρότερη περίπτωση κάποιον ε, ο οποίος είναι φορέας μιας νέας ιδεολογίας η εικόνα για ένα ταξίδι στο φεγγάρι όπως αυτό το οποίο περιέγραψε η κυρία Φοντελάιν ίσως δεν είναι εντελώς ε, άστοχο. Μετά την ε, έκρηξη μιας δεξαμενής ε, οξυγόνου, οι αστροναύτες δεν μπορούσαν να κάνουν απολύτως τίποτα. Ο ίδιος κίνδυνος απειλεί και τη συμφωνία της κυρίας Φοντερ Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών, εκ μέρους του ECR, για 1,5 λεπτό ο κύριο Μπουρζουά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει να είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει γεωπολιτική, να δημιουργήσει θέσει απασχόληση, να δημιουργήσει ευημερία, να φροντίσει κατά τη κλιματική αλλαγή και αναρωτιέται κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτές τις φιλοδοξίες η ε, νέα ε, πράσινη συμφωνία. Ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή, στην, σε μια κλειστή αγορά που υπήρχε μέχρι τώρα, θα υπάρξει πρόσβαση με πολλές θέσεις απασχόλησης ε, σε όλες τις χώρες μας. Η συμφωνία αυτή θα είναι επίσης μια βιώσιμη συμφωνία η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται και αποτελεί μέρος της συμφωνίας Μερκοσούρ. Υπάρχει επίσης, υπάρχουν διάφορες αρχές που έχουμε και εμείς και που θα πρέπει και αυτές οι χώρες να τηρούν τις προδιαγραφές δηλαδή τις δικές μας πρέπει να τις έχουν και εκείνοι. Πρόκειται για, μια, για ένα διακανονισμό έξυπνο. Φτάσαμε σε αυτόν μετά από πολλές προσπάθειες, πολύ διάλογο και προβλέπονται μάλιστα και κυρώσεις στην περίπτωση που δεν τηρούν τις προδιαγραφές οι εταίρεις μας. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα υπάρξει διάλογο και μετά κυρώσει. Οπότε, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πούμε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι κακή καθόλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, για 1,5 λεπτό, ο κ. Σόλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και 20 χρόνια η συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση. Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Μια παροχημένη εντολή ε, προς την ε, Επιτροπή χωρίς καμία απολύτως ε, συμβολή του Κοινοβουλίου. Οι διαφορετικές προτεραιότητες οι οποίες έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια, τα κεφάλαια για τη βιωσιμότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος, και κοινωνικά θέματα δεν περιλαμβάνονται. Λίγες μέρες μετά την COP25 θέτουμε το εξής ερώτημα. Η συμφωνία αυτή είναι συμβατή με το Green Deal που έχει εξαγγείλει η πρόεδρος της Επιτροπής. Ε, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι, μόνο ένα παράδειγμα, δεν έχουμε χρόνο. Ο στόχος 13 η χώρα με τα μεγαλύτερα τροπικά δάση στον κόσμο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Και το ίδιο κάνουν και πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία Mercosur συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη καταστροφή των τροπικών δασών του Αμαζονίου υπέρ της συνέχισης καλλιεργιών στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν εσεί η Επιτροπή θέλετε να έχετε την προστασία του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα, ε, θα πρέπει να υπάρχει μια νομική δεσμευτικότητα όσον αφορά την κλιματική προστασία. Και αυτό αποσιάζει από αυτή τη συμφωνία καθώς και το ζήτημα της ε, βιωσιμότητας των ε, μεθόδων παραγωγής. Γι' αυτό θα πρέπει να διακόψετε εδώ την σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστούμε. για 1,5 λεπτό κύριε Μπεγκίν για τους μη γεγραμμένου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. 906 εκατομμύρια εκτάρια του Αμαζονίου χάθηκαν το 2019 και είναι ένα τρίτο του, του Βελγίου που κάει και σε λίγου μήνε. Δεν ξέρω ποιε άλλε αποδείξει χρειάζονται για να αποδείξουμε τη συμφωνία με τι χώρε τη Λατινική Αμερική θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι πυρκαγιέ που είδαμε το καλοκαίρι και που συνεχίζουν μέχρι σήμερα ε, δημιουργούν ε, νέο έδαφο ή καλλιέργειε, κυρίω βοσκότοπου. 80% ε, είναι υπεύθυνοι για την αποδάσωση του Αμαζονίου. Η αποδάσωση δεν είναι το μόνο πρόβλημα το περιβαλλοντικό τη συμφωνία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν όρια συγκεκριμένε καιρό όσον αφορά την χρήση παραστοκτόνων, την εκμετάλλευση των ε, ηχθείων στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, η εκμετάλλευση των δετίνων πηγών όπω συμβαίνει στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Κατά την άποψή σα, αν αυτέ είναι οι ε, υποθέσει και οι βάσει, τι αποτελέσματα μπορεί να έχει μια συμφωνία, ώστε να μπορέσουμε να γίνει μεγαλύτερη εξαγωγή κρέατο και αγροτικών προϊόντων στην την Ευρώπη. Σε τι χρησιμεύει να λέμε στου παραγωγού μα να ρίπαν λιγότερο και να σέβονται πρότυπα ύψιστα όταν οι ανταγωνιστέ του στον κόσμο δεν πρέπει να σέβονται ούτε ένα από, μία από τι υποχρεώσει. Σε τι χρησιμεύει, περιορίζουμε τι εκπομπέ στην Ευρώπη, όταν οι πυρκαγιέ στην Αμαζονία παρήγαγαν 140 εκατομμύρια τόνου διοξιδίου του άνθρακο σε ένα μόνο καλοκαίρι. Συνάδελφοι, το περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα. Ο Αμαζόνιο είναι ο πνεύμονά μα. Και εμεί, εμεί πρώτοι θα πρέπει να προστατεύσουμε τον Αμαζόνιο. Αληθεύει το παγκόσμιο εμπόριο, δέχεται επίθεση και πρέπει να αντιδράσει μέσω συμφωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια συμφωνία όπω αυτή που έχουμε τώρα, εμεί δεν έχουμε πιστεί. Θέλουμε να δούμε περισσότερα χέγγια για του Ευρωπαίου καλλιεργητέ, ένα σχέδιο δράση για την προστασία του Αμαζονίου μέσω κυρώσεων που θα μπορούν να εφαρμόζονται με στόχο για, πολιτικ... για δεσμεύση των περιβάλλων. Είναι σημαντικό το εμπόριο να εμπορευόμαστε. Είναι ουσιαστικό. Η, Αμερική, η Λατινική είναι σημαντικό στρατηγικό εταίρο για την Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει εις βάρος των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος που είναι, ε, ανήκει σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, Επίτροπε Χόγκαν, με το νέο σας τίτλο που είσαστε ε, Επίτροπος για το Εμπόριο. Καλή τυχή για το μέλλον. Φύγατε, πήγατε από το τηγάνι, πηδήξατε στη φωτιά, θα έλεγα. Α, μεταξύ σφυρία και άκμονο είσαστε, διότι κανένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι εύκολο. Αυτό που συζητάμε σήμερα, συζητάμε δύο πράγματα που ακόμα δεν έχουν ζωντανέψει. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια συμφωνία που έχει επιτευχθεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί και μετά ο τίτλο με τρία λόγια που ακόμα δεν είδαμε τι λεπτομέρειε συμφωνία και ήδη πανικοβαλόμαστε. Θυμάμαι παλιά, όταν ο Πίτερ Μάντελσον ήταν υπεύθυνο για το εμπόριο, επίτροπο στη θέση σα και τότε οι Ιρλανδοί καλλιεργητέ ανησυχούσαν ιδιαίτερα για δίποτε προοπτική εμπορική συμφωνία. Οπότε γνωρίζετε ακριβώς τι θέλω να πω. Θα ήταν επικοδομητικό αν μας δίνατε κάποιες διαβεβαιώσεις σχετικά με το αντίκτυπο πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία θα έχει επί των Ευρωπαίων καλλιεργητών. Θα υπάρξει μείωση όσον αφορά την παραγωγή κρέατος εντός της Ευρώπης για να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση της εμπορικής συμφωνίας, της απαιτής εμπορικής συμφωνίας και αν η διαθέτηση είναι καλή ή κακή. Σήμερα το πρωί ένα ψήφισμα σχετικά με την προστασία των επικονιαστών και πώς να αποκατασταθεί η κατάστασή του. Και συζητήσαμε κυρίω τα, φυτο, τα προϊόντα φυτοπροστασία και τα παρασιτοκτόνα. Κάποιοι θέλανε να τα απαγορεύσουμε τελείω, άλλοι τα χρησιμοποιούμε λιγότερο. Δεν πάμε το κάνουμε αυτό όσον αφορά το Μερκοσούρ, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Και επανειλημμένα το συζητήσαμε αυτό και μα είπαν ότι υπάρχει αντιστοιχεία, ισοδυναμία. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε αυτή ε, τη συμφωνία, ισοδυναμία. Και πώ μπορούμε να εγγυηθούμε Πολύ καλά είπατε, καλά τα είπατε στην ομιλία σας. Αναφερθήκατε στο θάνατο του συμφωνίου στον φάτα περιβαλλοντικά. Πώς είμαστε σίγουροι ότι θα εφαρμοστούν οι σωστές συμφωνίες, ε, οι σωστές προδιαγραφές για το περιβάλλον στις συμφωνίες της χώρας Μερκοφούρ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Λάγκη έχει το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Το πλεονέκτημα αυτής της συζήτησης είναι ότι η συμφωνία Μέρκοσούρ δεν έχει ολοκληρωθεί και ε, ίσως θα υπογραφεί το 2021. Και βεβαίως ε, έχουμε χρόνο προκειμένου να εξελιχθεί περαιτέρω η συνθήκη, η συμφωνία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ορισμένα σημεία είναι διευκρίνιστα. Βέβαια υπάρχει ένα κεφάλαιο περί βιωσιμότητας, όπου η εφαρμογή ε, ε, που στήσαμε για την κλιματική αλλαγή τίθεται, καθώς και το ζήτημα ε, της βιώσιμης ε, γεωργίας. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κατά 60% περισσότερη αποψήλωση των δασών με το Μπολσονάρο και εγκρίνονται όλο και περισσότερα φυτοφάρμακα που είναι στην Ευρώπη απαγορευμένα. Επίσης δεν ε, κατοχυρώνεται η γη των αυτοχθόνων πληθυσμών. Και διαπιστώνεται μια παραβίαση, κατάφορη παραβίαση πολλών ε, κανόνων. Το ζητούμενο δεν μπορεί παρά να είναι τρία πράγματα. Πρώτον, χρειαζόμαστε συστήματα παρακολούθησης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν γίνονται αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα από αυτές τις αποψηλωμένες περιοχές. Ε, θα πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, βιωσιμότητα, εδώ θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα εν σχέση με την ε, βιώσιμη δασοκομεία και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και τρίτον, Χρειάζονται επίσης ε, μηχανισμούς ε, που να λειτουργούν όσον αφορά την ε, διαφύλαξη των δασών. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Κάσμπρο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο αυτό το καλοκαίρι και η ρητορική της ηγεσία της Βραζιλίας για το κλίμα σίγουρα δημιούργησαν πάρα πολλές ανησυχίες για τη συμφωνία αυτή Μερκοσούρ. Αλλά ας ε, καθίσουμε ψύχρεμα να δούμε τα γεγονότα. Τι λέει αυτή η συμφωνία. Στην πραγματικότητα η συμφωνία αυτή θα καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική τη Συμφωνία των Παρισιών, όχι λιγότερο, γιατί τελικά λαμβάνεται υπόψη το κλίμα στις εμπορικές μας συμφωνίες. Φιλόδοξα μέτρα πρέπει να λυθούν για να σωθεί το κλίμα πρέπει να τηρήσουμε τις συμφωνίες των Παρισίων, αλλά αυτό δεν θα το πετύχουμε αν δεν το κάνουμε μαζί με τους άλλους. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για μας συνεργασίας, για να πιέσουμε και να δημιουργήσουμε κίνητρα, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι μας να αναλάβουν τις ευθύνε τους. Περισσότερες εμπορικές συμφωνίες με δεσμευτικά κεφάλαια όσον αφορά τη βιωσιμότητα είναι αυτό που θα ευνοήσει την παγκόσμια συνεργασία. Οπότε να χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο τις εμπορικές συμφωνίες για να σώσουμε το κλίμα, αντί να τι αντιμετωπίζουμε σαν να πρόκειται για εχθρού του κλίματο. Θα μπορέσουμε, εφόσον υπάρχει καλύτερο νομικό πλαίσιο, να πετύχουμε περισσότερα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Μπρικμόντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Συμφωνία Ευρώπης Μερκοσούρ είναι συμβατή με τις φιλοδοξίες της Green Deal. Ναι, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Άρα όλε οι εμπορικέ συμφωνίε πρέπει να είναι συμβατέ με τι συμφωνίε του Παρισιού. Πώ όμω μπορούμε να πετύχουμε το 2050 με ιδανικό διοξίδιο του άνθρακα, όταν έχουμε από την άλλη μεριά τέτοιε χώρε. Τι θα γίνει με το διοξίδιο του άνθρακα. Ξέρετε ότι στη Γεωργία και μόνο οι εκπομπέ επιπλέον διοξιδίου του άνθρακα που ε, θα προσθεθούν ε, σε αυτές των Βρυξελών θα είναι ακριβώ αυτές. Και στη Μαδρίτη φάνηκε ότι η Βραζιλία θέλει να εμποδίσει μια φιλόδοξη συμφωνία. Συνεπώ, η συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ δεν φαίνεται να βελτιώσει τα πράγματα παρά το σαλέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πράσινη Συμφωνία λέει ότι όλοι οι κλάδοι πρέπει να συνεισφέρουν, όλοι οι τομεί. Κι όμω υπάρχει το γεωρικό μοντέλο και η εμπορική μας πολιτική που μας εμποδίζουν να καταλήξουμε στις συμφωνίες αυτές όπως είναι αυτή του Green Deal είναι μια δοκιμή η συμφωνία αυτή με τη Μερκοσούρ για το κατά πόσο μπορούμε να πετύχουμε τόσα λέει Πράσινη Συμφωνία. Αν επικυρωθεί μια τέτοια συμφωνία όπως είναι η Μερκοσούρ δεν θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Μάντισον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία Μερκοσούρ θα οδηγεί σημαντική αύξηση εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση τοποιημένο προϊόντων δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στον φάρο αγροτικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζει ένα φλεγωμένο κρίση περαιτέρω. Επίση, θα συμβάλλει στην ε, αγροτική κρίση σε πολλέ χώρε, όπω στη χώρα μου στην Εστονία. Και Εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για να μεταφορφωθεί η ευρωπαϊκή κοινωνία για να πετύχει ουδετερότητα για τον άνθρακα μέχρι το 2050. Οι χώρε όπως η Κίνα και η Ινδία δεν έχουν τέτοιο περιορισμό και αναπτύσσουν τι οικονομίε τους. Η Νέα Πράσινη Συμφωνία θα είναι ει βάρο των πλέον πολύτιμων μελών τη κοινωνία μας, εκείνων που μα δίνουν τρόφιμα, εναντίον των γεωργών μα. Η Πράσινη Συμφωνία θα έχει επιπτώσει στον αγροτικό τομέα, αλλά και χώρε που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα για την ενέργεια. Και σαν αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι που ζουν από αυτού του τομεί θα επηρεαστούν. Εστονία, παράδειγμα, είναι αυτάρκης όσον αφορά την ενέργεια. Βασίζεται όμω στα αποθέματα πετρελαίου τα δικά τη γι' αυτό. Με την έπαρση συμφωνία, η Εστονία θα υποχρεωθεί να βασιστεί σε άλλε χώρε για την ενέργεια. Αυτό με τη σειρά του θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα τη χώρα, την ανεξαρτησία τη και την κυριαρχία τη. Πιο σοβαρό αυτό. Οι εναλλακτικέ μορφέ ε, ενέργεια θα βρισκόταν στα βιοκαύσιμα, υποτίθεται. Σύμφωνα πρόσφατα πορίσματα για την πείνα και την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα βιοκαύσιμα αποτελούν λύση. Πιθανότατα θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Λόγω φυσική, φυσικών νόμων, οι ποιότητε των βιοκαυσίων που χρειάζονται για την παραγωγή ενέργεια, αυξάνουν τα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Εάν σπαταλάμε, σπαταλάμε ενέργεια για να παράξουμε ενέργεια και γη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να παράξει τρόφιμα, παράγεται ανταυτού για την παραγωγή ενέργεια. Και αντί να μιλάμε η συμβατότητα τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώσεω Μερκοσούρ με τη Πράσινη Συμφωνία, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για την καταστροφικό αντίκτυπο που θα, είχε, θα είχαν οι πρωτοβουλίε για του γεωργού συγκεκριμένα και του Ευρωπαίου πολίτε εν γέννη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο ομιλητή για ένα, λεπτό, κυρία Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρώπη συζητάμε έτσι πολύ της μόδας για την Πράσινη Συμφωνία και μετά φαίνεται η υποκρισία μιας συζήτησης που ενώ έχουμε και βάζουμε νέε υποχρεώσει στους αγρότε, από την άλλη μεριά μειώνουμε τι υποχρεώσει για τα εισαγόμενα. Το πρόβλημα είναι ότι τα προϊόντα αυτά και τα δικά μα και τα εισαγόμενα ε, βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ένα παγκόσμιο χώρο χωρί όμω ίδιους κανόνε. Εμεί βάζουμε όλο και περισσότερου κανόνε για το περιβάλλον. Στην Περκοσούρ, όμω επιτρέπονται τα αντιβιωτικά με ορμόνε αυξητικέ και γενετικά τροποποιημένα. Οπότε πρέπει να επιθυμησουμε τι αυστηρέ προδιαγραφέ που οφείλουν να έχουν οι δικοί μας αγρότες σε θέματα φυτογειονομικά και για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Όσα αναφέρονται όμως για τη βιωσιμότητα στη Συμφωνία Μερκασούρ πρόκειται απλώς για δήλωση προθέσεων και ξέρουμε πώς παράγουν τα τρόφιμά τους στη Μερκοσούρ. Οπότε τίθεται σε κίνδυνο και η παραγωγική δύναμη των δικών μας χωρών, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και συνέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για πράσινη συμφωνία και για βιώσιμη γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μορέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο το νέο Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο συνάδει με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Ε, για μένα η απάντηση είναι προφανώς όχι. Και πραγματικά εκπλήσωμε, αλλά σχεδόν θα έλεγα θαυμάζω του συναδέλφου τη δεξιά που μα εξηγούν ενθουσιαστικά ότι χάρη σε αυτή τη συμφωνία ο κ. Μπολσονάρο θα μεταμορφωθεί θαυματουργά σε προασπιστή του περιβάλλοντο και των αυτοχθόνων πληθυσμών. Αγαπητέ συνάδελφοι, αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία όχι δεν συνάδει. Καταρχά, διότι τίποτα παρά τη αύξηση των ποσοστών των εξαγωγών τη όγια, για εθανόλη, για το βόη, για τα πουλερικά, για τη ζάχαρη, αντιπροσωπεύουν 9 εκατομμύρια τόνου παραπάνω για τα αερίου του θερμοκηπίου. Όχι, δεν συνάδει, δεν είναι συμβατό με, με, το Πράσινο Σύμφωνο, διότι οι φίλοι τη αγροτοφομικού τομέα του κ. Μπολσονάρο εξακολουθούν να καταστρέφουν τον Αμαζόνιο. 93% συμπληρωματικών πυρκαγιών φρέτο, πρόσθετων πυρκαγιών. Όταν διαβάζουμε ε, το κείμενο, η αρχή τη πρόληψη αποδυναμώνεται και θα εκτεθεί η Ευρώπη σε όλο και περισσότερο επικίνδυνα προϊόντα. Βλέπαμε το COP25 στη Μαδρίτη τι έγινε, ότι η Βραζιλία μαζί με άλλε χώρε εξάλλου ασταμάτητα αμφισβητούσαν κάθε προάσπιση αρχή τη πρόληψη των Ευρωπαίων. Σίγουρα αυτό δεν είναι συμβατό, αυτή η συμφωνία δεν συμβατή και μην είστε αφελεί ή μην είστε υποκριτικοί τουλάχιστον. Υποκριτέ, συγγνώμη. Τουλάχιστον ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή για 1,5 λεπτό, ο κύριο Σίντσιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει με τάχιστο ρυθμό και οι πολιτικές που βασίζονται στη βία δεν μπορεί να πετύχουν η, εξαιρετική, η, αλλαγή του κλίματος και οι ακραίες συνθήκες του κλίματος ακούστηκαν και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ακούστηκαν και ζητηθήκαν αυτά. Η, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που συνέβαιναν μια φορά κάθε 100 χρόνια τώρα μπορούν να συμβαίνουν κάθε χρόνο. Από το 1970 μέχρι σήμερα εμείς σαν άνθρωποι σκοτώσαμε 60% όλων των ζώων που υπήρχαν στον κόσμο. Και είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να καταστρέφουμε και τα έντομα. Το συζητήσαμε αυτό χθε στο κάτω-κάτω. Από... πότε, μέχρι πότε θα είμαστε τόσο υπερφύαλοι και μέχρι πότε θα είμαστε έτσι χωρίς να σεβόμαστε το περιβάλλον. Στην αρχή του 21ου αιώνα δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε επί των πολιτικών του 20ου ή του 19ου αιώνα για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τον Αμαζόνιο και τα δάση του Αμαζονίου, τα τροπικά δάση, θα πρέπει να αντιταχθούμε στον ειδονισμό, θα πρέπει να αντιταχθούμε στη βία, θα πρέπει όλα αυτά να τα παρνηθούμε. Ε, ε, έχει γίνει πάρα πολλή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν τεράστια χρέη και θα πρέπει να εξετάζουμε τα θέματα σε μεγαλύτερο βάθος και δεν θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό, κύριος Γκαρσία Μαργάγιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε μπροστά μας ένα δίλημα. Ή ελεύθερο εμπόριο ή προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη γνώμη μου όμως δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Οι ακροφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή ή ότι η κλιματική αλλαγή δεν οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Οπότε οποιαδήποτε συμφωνία εμπορική, είτε προβλέπει είτε δεν προβλέπει επιφυλάξεις, δεν έχει καμία σημασία. Οι άλλοι πάλι πιστεύουν ότι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία είναι ένα κόλπο για να μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει για το περιβάλλον και βάζω τον Πολσονάρο σαν παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου το δίλημα αυτό είναι ψεύτικο. Πρέπει να προσαρμόσουμε την προσαρμογή του περιβάλλοντος με το άνοιγμα των συνόρων για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου η συμφωνία αυτή το καταφέρνει αρκετά καλά γιατί λέει συμφωνία ότι γίνονται σεβαστές όλε οι συμφωνίε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ότι πρέπει να υλοποιηθεί η συμφωνία των Παρισίων που αποφεύγει την ε, αποψήλωση και προστατεύει τα δάση. Επίσης, προβλέπεται κοινωνική ευθύνη των ιδιωτικών επιχειρήσεων και επίσης γίνεται και μνήμα για το πώς λύνονται οι διαφορές, με συγκεκριμένους κανόνες επίσης για τη διατροφική ασφάλεια. Οπότε η ομάδα μου είναι υπέρ της συμφωνίας αυτής με τη Μερκοσούρ, γιατί πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή σέβεται τις δεσμεύσεις που έχουμε ε, αναλάβει μέσα στην Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία υπέρ του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε δύο λεπτά τώρα. Γκούτελαντ. Θα περιμένουμε την κυρία Κούτελαντ. The floor is yours, please. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λυπούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία επιτέλους ε, ε, βρίσκεται καθοδόν και υπάρχει μια στρατηγική προκειμένου να προωθηθεί μια δομική ε, αναδιάρθρωση. Και πράγματι πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία με το Green ε, Deal. Συγγνώμη που είμαι λαχανιασμένη, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να πάρω το λόγο και είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτή η πράσινη συμφωνία συνδέεται με πολύ υψηλές προσδοκίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας αποδείξει ότι είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει το θέμα αυτό σε όλους τους πολιτικούς τομείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πακριβώς την υφιστάμενη νομοθεσία. Εμείς από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών επιθυμούμε αυτή τη μεταβολή για ολόκληρη την Ευρώπη και ελπίζω ότι η νέα γενιά η οποία διαδελώνει στους δρόμους της Ευρώπης έχει την αίσθηση ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις, ε, τα αιτήματά της και ότι θα δεσμευτούμε για μια αλλαγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Green Deal σημαίνει ότι εννοούμε σοβαρά ένα βιώσιμο μέλλον και ε, με αυτά τα θετικά λόγια έναντι της Επιτροπής ε, θα ήθελα να πω ότι από την άλλη ε, το Green Deal ε, συνιστά και μια δέσμευση βεβαίως. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι να στρώσουμε ένα κόκκινο χαλί για το Green Deal αλλά απαιτείται ένα συνεχή ε, διάλογο επί τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα πρέπει να μα προβληματίσουν αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά το έργο μα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ε, να στρέψουμε τη ματιά μας προς το μέλλον και να έχουμε ξεκάθαρα κατά νου ότι εμείς ε, ως ε, ηγετική ε, δύναμη θα μεριμνήσουμε γι' αυτά. Ε, όσον αφορά τη διάσκεψη της Γλασκόβης, το, η Πράσινη Συμφωνία είναι κάτι που έχουμε στα χέρια μας, αλλά στη βάση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη την προετοιμασία των εργασιών στη Γλασκόβη, ούτε ώστε όλες οι χώρες να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου μια ξεκάθαρη στρατηγική. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Ραφαέλα. Κύριε Πίτροπε, οι πρόσφατε εξελίξει στον ΠΟΕ μα έδειξαν πόσο πολύτιμο είναι το ότι η Ευρώπη έχει αυξανόμενη συνεργασία με τρίτε χώρε. Δεν χρειάζεται κανεί να είναι διάνοια για να δει πόσο καλό είναι να έχει κανεί πλήρε εμπορικέ σχέσει με Ιαπωνία, Καναδά, Σιγκαπούρη και πολλού άλλου. Όπω και άλλοι, ε, καταστρέφουν αυτά που είχαν ε, δημιουργηθεί επί δεκαετίες. Θα πρέπει αυτές οι συμφωνίες να γίνουν όσο το καλύτερο γίνεται βάσει των αξιών μας και με σεβασμό του περιβάλλοντος. Πώ θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι χώρε τη Μερκοσούρ θα σεβαστούν τη Συμφωνία των Παρισίων. Και αν όχι, ποιε θα είναι οι συνέπειε. Η Ευρώπη τα κατάφερνε καλύτερα όταν χρησιμοποιούσε την οικονομική τη δύναμη για το καλό στον κόσμο, με περαιτέρω εργαλεία και αποτελεσματικότερη επιβολή, όπω αυτά αναφέρονται στην Πράσινη Συμφωνία, μπορούμε να κάνουμε βήματα προ σωστή κατεύθυνση. Και γι' αυτό το λόγο καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει πρακτικά την κανονισμό περιλωτομία για να σωθεί ο Αμαζόνιο που είναι κρίσιμο κομμάτι του παγκόσμιου οικοσυστήματό μα και πατρίδα των ηθαγενών πληθυσμών, των οποίων τα θεμελιώδη δικαιώματα απειλούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα, για ένα λεπτό, η κυρία Τσάουνς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, το κεντρικό ερώτημα είναι η συνέπεια. Η εμπορική μας πολιτική είναι συνεπής, συνάδει με τους στόχους για το κλίμα. Σε σχέση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσης Μερκοσούρη, η απάντηση είναι ουχή. Βεβαίω, αληθεύει ότι το εμπόριο μπορεί να υποφελές και για τα δύο μέρη. Κάθε παιδί μπορεί να σα πει ότι η ανταλλαγή καρτών μπορεί να γίνει μεταξύ παιδιών και είναι ε, χρήσιμη, αλλά δεν είναι καλό κάθε είδους εμπόριο. Και το ούτω αποκαλούμενο εμπόριο, ε, ελεύθερο εμπόριο έχει οικολογικό και κοινωνικό κόστο. Όλοι έχουμε πληρώσει το τίμημα για την καταστροφή των δασών και για την αλλαγή του κλίματο. Η εξαγωγή περισσότερων αυτοκινήτων ορυχτών καυσίμων από την Ευρώπη και να δεχόμαστε περισσότερο βόλιο κρέα από εκεί που εκτρέφεται σε πρώην δάση του Αμαζονίου δεν είναι κάτι καλό. Επίτροπε, επίτροπε ε, Χόγκαν, ε, προ, ε, Υπουργέ ναι. ε, είπατε ότι χρειαζόμαστε στεναρή πολιτική. Δεν είναι ανόητο το περιεχόμενο. Να, να πούμε πιο ξεκάθαρα στα σχετικά κεφάλαια, δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο τροχοπέδι στον κύριο Μπολσινάρου. Αναφερθήκατε στη δέσμευση στο άρθρο 5. Αλλά ο πρόεδρος Μπολσονάρο ειλικρινά δεν Σκασίλα του για τον Αμαζόνιο, σκασίλα του για το κλίμα. Είδαμε πόσο καταστροφικά ήταν τα αποτελέσματα στην COP25 την προηγούμενη φορά. Κάποιοι συνάδελφοι αλλού στο Κοινοβούλιο είπαν ότι θα έχουμε μεγαλύτερη μόχλευση αν υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο ότι αυτό συμβαίνει. Το σημείο τη μόχλευση είναι πριν υπογράψουμε. Χρειαζόμαστε αποδείξει συγκεκριμένη αλλαγή και βελτίωση στοιχεία επίση και από τη δική μα πλευρά ότι η εμπορική πολιτική μα ταιριάζει με του στόχου για το κλίμα και τη επικοινότητα. Σα καλώ να το εξασφαλίσετε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή για δύο λεπτά, ο κύριο Λαντσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ είναι από τι σημαντικότερε εμπορικέ συμφωνίε που μπορεί να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 780 εκατομμύρια ανθρώπου. Ε, παρά το γεγονό αυτό, σήμερα ε, βλέπουμε συνολικά τι εμπορικέ συμφωνίε, μεταξύ των οποίων και αυτή με το Βιετνάμ, και κατά πόσον συνάδουν με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά μα πρότυπα. Θα πρέπει όλε οι δημοτεύσει να λάβουν υπόψη τα ειδικά συμφέροντα των διαφορών τομέων και να υπάρξει αρχή τη αμοιβαιότητα. Όχι να θυσιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δώσουμε ε, σε ορισμένου παραγωγικού κλάδου την προτεραιότητα σε αντίθεση με άλλου και όπω συνήθω ει βάρο του περιβάλλοντο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για αυστηρή παρακολούθηση τη υλοποίηση τη συμφωνία. Όμω εδώ παραμένουν πολλέ ανησυχίε, όχι μόνο για το τι θα γίνει με το λιγμένο βόλιο κρέα, αλλά και με την ε, μεταποιητική βιομηχανία των χωρών ε, τη περιοχή του Μερκοσούρ και ε, το δεδομένο των αυστηρών προτύπων που επιβάλλουμε εμεί στι χώρε μα. υπάρχουν φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στο Μερκοσούρ, τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και η εκτροφή πουλερικών είναι από αυτέ που είχαν απαγορευτεί ω μέθοδο εκτροφή στην Ιταλία το 2018. Μετά για τη ζάχαρη, το ρύζι και για τα ε, Υπάρχουν φυτογενομικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με παράσιτα τα οποία ε, είναι διαδεδομένα στην ε, Νότια Αμερική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, ότι η διαφιλονικία με την κυβέρνηση τη Βραζιλία έχει, έχει έρθει στο επίκεντρο τη προσοχή αντί να ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα στι συμφωνίε αυτέ που δεν πρέπει να βρίσκονται σε δεύτερη θέση. Και να υπάρχει έλλειμμα για την προστασία του περιβάλλοντο. Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα των χωρών με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι συνεπή με τι ε, τόσο συχνά ε, ανακηρυγμένε ε, υπέρτατε αρχέ τη περιβαλλοντική προστασία, θα πρέπει να επιβάλλουμε την, ε, χρήση την ε, παραγωγή πλαστικών μια χρήση και στι χώρε με τι οποίε έχουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Διότι οι βάλλο πληρώνουν πάντοτε το τίμημα Ευρωπαίοι πολίτε και ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Ο κύριο Ράισεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Και σήμερα στην Ολλανδία έχουμε πάλι διαμαρτυρίες γεωργών και το καταλαβαίνω πολύ καλά, διότι οι γεωργοί είναι στριμωγμένοι. Από τη μια έχουν ένα πλήθος κανόνων και από την άλλη πολύ μικρά περιθώρια. Και συνεχώς τους ταπεινώνουν. Και χτες ε, ο συνάδελφός σας Τίμερμανς, ο οποίος τους θεωρεί άνθρωποι που είναι ε, αγκιστρωμένοι σε απαρχιωμένες ιδέες. Πώς έτσι, απαρχιωμένες. Η Ευρώπη προχωράει, τρέχει. Αυτό θα πρέπει να το αντέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βλέπω την πράσινη συμφωνία, είναι τεράστιες οι φιλοδοξίες και μηδέν ρεαλισμός. Πολύ ψηλή στόχη και καθόλου εργαλεία για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Για ποιο λόγο διαρκεί τόσο πολύ η έγκριση να κυκλοφορούν νέα φυτοφάρμακα πράσινα και συνεχίζουμε τις φθηνές αγωγές από τη Μερκοσούρ που όπου υπάρχουν τελείως διαφορετικοί κανόνες. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα για μας. Αυτό που ζητώ είναι ε, πραγματική περηφάνεια για όσα έχουν γίνει, όπως τους αρμόζει, ρεαλισμό και ίσους κανόνες παιχνιδιού. Μόνο έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε προς την βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Ουρμπάν Κρέσπο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μπολσονάρο είπε ότι η Βραζιλία αποχωρεί από τη Συμφωνία των Παρισίων και θα συνεχίσει να αποψηλώνει τον Αμαζόνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανήγγειλε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει εμπορικέ συμφωνίε με χώρε που δεν θα κυρώσουν τη συμφωνία για το κλίμα. Πριν από λίγε εβδομάδε το Κοινοβούλιο ε, κήρυξε κατάσταση έκτακτη ανάγκη για το κλίμα και πριν από λίγε μέρε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταβαίων και Κλάδων κατέβασε τη νέα πράσινη συμφωνία. Όλα αυτά είναι άκυρα όταν μιλάμε για εμπόριο στην υπηρεσία των πολιεθνικών. Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με την μισόγυνη ακροδεξιά κυβέρνηση ε, του Μπολσονάρ και με το Μερκοσούρ. Άλλη μια υποκρισία που διέπει ε, την ε, οικονομική πολιτική. Πώς μπορείς να κηρύσεις έκτακτη ανάγκη για το κλίμα και να υπογράφεις συμφωνίες που καταστρέφουν τα δάση από τις εξορρυκτικές και τις εντατικές αγροτικές δραστηριότητες. Και είναι καταδικασμένοι οι ακτιβιστές και ακριβίστριες στην Βραζιλία, όπως ε, μας έδειξαν σήμερα οι φιναλίστ του βραβείου Ζαχάροφ. Αν η ερώτηση είναι αν αυτή η συμφωνία Μερκοσούρ είναι συμβατή με τη νέα πράσινη συμφωνία, η απάντηση είναι αρνητική. Όχι. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και να καταρρύψουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπούντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι. Οι εμπορικές ε, συμφωνίες είναι απαραίτητες για οποιαδήποτε σοβαρή εμπορική δραστηριότητα. Από την πλευρά όμω των αγροτών το να μιλάμε για τη συμβατότητα μεταξύ της Συμφωνίας Μερκοσούρ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δεν έχει νόημα. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Είναι διπλά τα στάνταρτ. Καταρχάς, ε, η πάταξη της κλιματικής αλλαγής. Είναι περίπλοκο να μιλάμε για βιωσιμότητα των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δίνουμε σοβαρά κονδύλια γι' αυτό. Ενώ στο Μερκοσούρ οι χώρες και τα δάση τους ε, με πρόθεση για να φτιάξουν χώρο για άλλα προϊόντα. Επίση, μιλάμε για το Farm to Fork ω στρατηγική. Θέλουμε υψηλά στάνταρ για όλα τα προϊόντα. Όλα τα τρόφιμα που παράγονται από του αγρότε στην Ευρώπη, ενώ στι χώρε τη Μερκοστούρ δεν υπάρχουν τέτοια στάνταρ. Επίση, έχουμε εισαγωγέ σε ε, βόλου κρέατος από την Βραζιλία και δεν μπορούν οι Ευρωπαϊκέ Υπηρεσίε να το ανοιχνεύσουν. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Και ε, επίσης οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίως ε, έχουν, ε, το, έχουν την υποχρέωση να σέβονται διατάξεις για τις ορμόνες και τα λοιπά όταν οι αγρότες στη Μερκοσούρ δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Θέλουμε λοιπόν ξεκάθαρες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα για να διασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των αγροτών στο Μερκοσούρ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο για 1,5 λεπτό είναι ο επόμενος ε, ομιλητής. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Χόγκαν, με την Πράσινη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνάψει ένα νέο σύμφωνο για τους πολίτες και τους καταναλωτές της. Ένα σύμφωνο που χάρη στην στρατηγική που τώρα συζητάμε μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω και να στραφεί προς την ποιότητα των τροφίμων ε, και από την σκοπιά του προϊόντος, του τελικού προϊόντος που θα πρέπει να είναι υγιές και από την σκοπιά της ισότιμης, βιώσιμης και διαφανούς ε, μεθόδου παραγωγής. Η παραγωγή της Ευρώπης, ε, αγρότες και κοινοτρόφοι, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση ενισχύοντα τα παραγωγικά μας πρότυπα. και Είμαστε ούτω ή άλλω μεταξύ των πιο προηγμένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να του εγκαταλείψουμε μόνο του. Θα πρέπει μάλιστα να δώσουμε έμφαση στι προσπάθειέ του αντιμετωπίζοντα όλε τι υποθέσει αθέμετου ανταγωνισμού ε, σε σχέση με παραγωγού τρίτων χωρών. Πρόκειται για έναν στόχο, τον οποίο δεν μπορούμε πλέον να παραβλέπουμε, κύριε Επίτροπε, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην ε, προτινόμενη συμφωνία για τις χώρες Μερκοσούρ. Η επισητιστική διπλωματία τη Ευρώπη είναι πολύ σημαντική πλέον και θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των εμπορικών μα εταίρων. Πρέπει να γίνουμε πραγματικά σημεία αναφορά σε διεθνέ επίπεδο. Με ορισμό των αγροτικών, κτηνοτροφικών και επιστημιστικών προτύπων παραγωγή. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κύριο Yeah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ ε, θα είναι ωφέλιμη για όλους μας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όμως δεν πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός, πρέπει να είναι το μέσο για κάτι άλλο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το τι συμβαίνει στη Βραζιλία με τις δασικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο. Πρέπει όλοι μαζί να μιλήσουμε για τα κλιματικά θέματα και να ασχίσουμε πίεση στον Μπολσονάρο ο οποίο χρειάζεται την συμφωνία του Μερκοσούρ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, περισσότερο και από εμά. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει το κλίμα, αλλά τον ενδιαφέρει μια ισχυρότερη οικονομία. Θα είναι τεράστιο πολιτικό σφάλμα, λοιπόν, μετά από 20 χρόνια σκληρή δουλειά ε, για αυτή τη συμφωνία να χαθεί σε ένα τέτοιο ε, παιχνίδι ε, και καλό θα ήταν να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση